neither reciprocity or a level playing field, so EU investors' access on Chinese markets still faces significant obstacles. That would be in one minute, but please read the report. It's a very interesting read. Thank you very much. Dankeschön. Und damit kommen wir jetzt, schließe den Tagesordnungspunkt 10 und kommen wir zu Punkt 11 unserer ersten, ja, ja, unserer ersten Abstimmung um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 Καλησπέρα σας. Να σας πούμε με χαρά ότι και πάλι αν χρειάζεται μπορείτε να ακούσετε την ελληνική διερμηνία στο κανάλι 7. Οι διερμηνείς σας εύχονται καλημέρα και ξεκινάμε. Οι Μεξικανοί λοιπόν θέλουν να συμφωνήσουν μαζί μας, θέλουν να επεκταθούμε σε νέους χώρους και όταν συζητά κανείς την πνευματική ιδιοκτησία, ίσως έφτασε η στιγμή να αρπάξουμε την ευκαιρία, οπότε το μήνυμά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασφανούμε α, εξίσου φιλόδοξοι και να ακούσουμε βεβαίως και τα ζητήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά Ας μην ξεχνάμε πως το δυναμικό για την Ευρώπη και, και οι ευκαιρίες είναι τεράστιες. Ας τις χρησιμοποιήσουμε και να δείξουμε και στην υπόλοιπη οικουμένη πως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δουλειές με όλους. Το Μεξικό άλλωστε είναι και η πύλη προς τη Λατινική Αμερική, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει εκεί να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Κύριο Σαλαβράγκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την επίσκεψη, αλλά άκουσα πως ε, η αποστολή αυτή πήγε πολύ καλά, με πολλά θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω πως είναι πολύ ε, δραστήριος εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμφωνία ε, σύνδεσης, μία από τις πρώτες συμφωνίες τέταρτης γενιάς που έδωσε πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα επίσης να πω πως αυτή τη στιγμή περνάμε σε μία φάση εξυγχρονισμού και ανανέωσης της τρέχουσας συνθήκης συμφωνίας και πιστεύω πως το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό του timing, δηλαδή καθυστερούμε. Στην Ολομέλεια ψηφίσαμε τη συμφωνία με τον Καναδά πρόσφατα και οι διαπραγματεύσει εδώ έχουν περάσει 7 χρόνια και ακόμα είμαστε στη διαδικασία επικύρωση. Το Μεξικό είναι μια χώρα η οποία έκανε πολύ σημαντικέ συνταγματικέ μεταρρυθμίσει που ενδέχεται να προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά για το χρόνο που χρειάζεται η διαδικασία μας. Μας το είπε άλλωστε και η Επίτροπος για το Εμπόριο και θα πρέπει να μπορέσουμε, όπως είπε και ο εισηγητής, να κλείσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση πριν τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Ιούλιο του χρόνου και να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολιτική συγκυρία. Ξέρετε πως μετά την εκλογή του νέου Αμερικανικού, Αμερικανού Προέδρου έχει ε, διάφορα θέματα το Μεξικό και εμείς αντιμετωπίζουμε κάτι αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως λοιπόν θα ήταν ευκταίο να δούμε να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκ μέρου των 28 διαπραγματεύεται, αν μπορεί να παρουσιάσει ένα χρονικό ορίζοντα, ο οποίο ήταν και ρεαλιστικό, αλλά και θα ανταποκρίνεται και στι φιλοδοξίε που παρουσίασαν και ο εισηγητή και οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να λάβουμε του χρόνου υπόψη μα, μα επηρεάζουν. Η Επιτροπή Juncker. σε λιγότερο από δύο χρόνια ε, φτάνει στη λήξη της θητείας της, να προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα και να κλείσουμε ε, στην ίδια γραμμή με τις προτιμησιακές ε, συμφωνίες που έχουμε προκρίνει πρόσφατα. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα χρησιμοποιήσω την δυνατότητα να μιλήσω στη γλώσσα μου, αλλά θα πω κάποια λόγια στα αγγλικά. Στην αρχή, Νομίζω πως, ε, όπως είπε και ο συνάδελφος, η κανάλιση ήταν πολύ καλή και το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε ήταν κατάλληλο. Και να πω επίσης ότι εξεπλάγει ευχάριστα όταν είδα τη δυναμική και τις δυνατότητες που έχει το Μεξικό. Πόσο μάλιστα τώρα που προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη συμφωνία με το Μεξικό. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την θέληση να συνεργαστεί, θέλει να χτίσει τείχη, οι Μεξικάνοι όμως θέλουν να χτίσουν γέφυρες. Γέφυρες ε, που θα διασχίζουν τα ραγμένα νερά, θα διασχίζουν τον Ατλαντικό ωκεανό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε και να είμαστε ένας ε, κατάλληλος εταίρος. Όπως είπα και πριν, πρέπει να ε, συνδυάσουμε τις προσπάθειες αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης με το Μεξικό. Και αυτό είναι κάτι που ε, μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσες δυνατότητες και ευκαιρίες δηλαδή υπάρχουν. Το Μεξικό μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως η φιλοδοξία είναι ε, απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χαουταλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μόησα και τους υπόλοιπους συναδέλφους που μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της αποστολής τους. Πράγματι, οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μπορούμε να συνάψουμε μια συμφωνία με το Μεξικό. Είναι η κατάλληλη στιγμή και πιστεύω πως μπορούμε να είμαστε γρηγορότεροι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά Έχω δει ότι έχουν γίνει πολλέ παρόμοιε ασκήσει στο παρελθόν με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, για παράδειγμα, και έχουμε δει τα προβλήματα που προέκυψαν, έλλειψη διαφάνεια στη διαπραγματεύση κτλ. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των επιχειρήσεων και σε αυτά των πολιτών και τη κοινωνία των πολιτών για την προστασία των εργαζόμενων. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Μόησα, ότι χρειάζεται το κεφάλαιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς να είναι πολύ φιλόδοξο και επίσης ε, το κεφάλαιο που θα αφορά τις κυρώσεις να είναι εξίσου σημαντικό και αυστηρό. Θα μπορούσε αυτή η συμφωνία να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τις μελλοντικέ ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μελλοντικέ συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τις ε, Δυνατότητε που μας δίνουν τα διδάγματα που αντλήσαμε. Μπορούμε λοιπόν και στην περίπτωση του Μεξικού να το χρησιμοποιήσουμε. Το Μεξικό χαρακτηρίζεται από μεγάλα ποσοστά τιμωρησίας, πάνω από 90% και αυτό φυσικά σημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν ελάχιστες ε, εγγύησεις, ελάχιστη ασφάλεια. Χρειάζεται λοιπόν ε, αυτό να αντιμετωπιστεί, αλλά και ε, το αντίστροφο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δηλαδή να έχουν υποχρεώσεις και ε, μεταξύ άλλων της καταπολέμησης και της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει λοιπόν ένα τεράστιο έργο μπροστά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να είναι ταχύτατη, όσο και ε, στην προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια δεδομένων των παρελθυντικών εμπειριών μας. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο, τα δικαιώματα των εργαζομένων, για παράδειγμα, αλλά και τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Σίγουρα αυτά θα αποτελέσουν πρόκληση για το Μεξικό Γι' αυτό χρειάζεται ταχύτητα και από εσά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γιώργενσεν, πότε θα έχουμε προτάσεις, πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Μου δώσατε την ευκαιρία λοιπόν και σας ευχαριστώ να συνεισφέρω στη συζήτηση, να σας πω εν συντομία πως έχουμε καταγράψει με πολύ ενδιαφέρον τις εντυπώσεις που αποκομίσατε από το Μεξικό για μας η στιγμή της δικής σας επίσκεψης ήταν πραγματικά επίκαιρη γιατί ήταν σημαντικό να δείξουμε στο Μεξικό πως υπάρχει στήριξη, υπάρχει ενδιαφέρον κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και τι καλύτερο παρά μία ε, αποστολή της ίντα με εκπροσώπηση όλων των πολιτικών ομάδων να σας πω πως επίσης καταγράψαμε με ιδιαίτερη προσοχή τη δική σας ε, ε, παρατήρηση πως θα πρέπει το περιεχόμενο να είναι το σωστό σε κάθε ε, κλάδο και σε κάθε κομμάτι της συμφωνίας. Έχετε δίκιο και η ανανέωση, η εξυγχρονισμό της συμφωνίας μας προσφέρει μια ευκαιρία να συμπεριλάβουμε μια σειρά από θέματα τα οποία δεν βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βοήθεια, αναπτυξιακή, ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα τα οποία μπορούμε να λύσουμε και στο πολιτικό σκέλος συμφωνίας. Τώρα, για τη διαφάνεια και την παρατήρηση που κάνετε εκεί, βεβαίως και θα το λάβουμε όντως υπόψη, νομίζω πως έχετε λάβει και τις εκθέσεις από τους γύρους διαπραγμάτευσης που έχουμε διεξάγει και έχετε δει επίσης και τα κείμενα ε, απογραφής ας πούμε και ελέγχου διαπραγματεύσεων που σας έχουμε δώσει ε, Τώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, αλλά όλα αυτά τα κείμενα θα σας τα καταθέσουμε ε, εν και του γύρου τον Απρίλιο. Ελπίζουμε ε, εμπρόθεσμα και πάντα ε, ε, είμαστε διαθέσιμοι για να έρθουμε να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα αυτά μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω και το λόγο στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Νομίζω κάπου κάθεστε. Ευχαριστώ. Είμαι ο επικεφαλής της μονάδας στην εξωτερική υπηρεσία δράσης για την Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική ε, και τα σχετικά θέματα και πρέπει να σας πω πως η κυρία Μογκερίνη είναι η αρμόδια που έχει την εντολή για την διαπραγμάτευση, την οποία έχει ε, παραδώσει στην, ε, στον Γενικό μας Διευθυντή και όπως και οι συνάδελφοι, έτσι και εμείς έχουμε καταγράψει τις συστάσεις σας και πιο συγκεκριμένα τη σύσταση για τον σεβασμό των βασικών αρχών που ε, μοιραζόμαστε με το Μεξικό στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό συμπεριλαμβάνει κοινωνικά και οικονομικά ε, δικαιώματα, όπως επίσης και την έκκλησή σας για διαφάνεια. Κάνουμε τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών για να τους ενημερώσουμε για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία και επειδή είναι μια ε, διαδικασία εν εξελίξει, όντως υπάρχουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ακόμα. Όμως με την κοινωνία των πολιτών μοιραζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις όταν θα φτάσει η στιγμή του να κλείσει η συμφωνία. Για το χρονικό ορίζοντα να σας πω πως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε όλα τα τμήματα του πολιτικού σκέλους της συμφωνίας τα έγγραφα χρειάζεται να υποβληθούν και στη σχετική ομάδα στο Συμβούλιο ε, που είναι για τις χώρες Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Και μόλις έχουν έχει καλός για το έγγραφο αυτό, θα το δώσουμε στους ε, Μεξικάνους ομολόγους μας, έτσι ώστε ελπίζω πριν το καλοκαίρι να έχουμε κλείσει τα περισσότερα από τα σημεία της συμφωνίας για να εξασφαλίσουμε πως η συμφωνία μπορεί να κλείσει και πριν τα τέλη της χρονιάς. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ελπίζω λοιπόν πως και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα συνεργαστούμε για μια καλή συμφωνία εν ευθέτω χρόνο. Παρεπιπτόντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την στήριξή σας στην αντιπροσωπεία μας στο Μεξικό. Πραγματικά είχε οργανωθεί πολύ καλά. Δεν ξέρω, ο συνάδελφος θέλει να κλείσει, ναι. Καταρχήν να σας πω πως το νέο σύστημα επίλυσης ε, επενδυτικών διαφορών που έχουμε δημιουργήσει για την ΣΕΤΑ και για την ΣΕΤΑ-ΣΥΝ ε, που έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Το νέο λοιπόν αυτό σύστημα αποτελεί και το σημείο θετηρίας για την όλη διαπραγμάτευση. Δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε οτιδήποτε που να προσεγγίζει το παλαιότερο σύστημα. Ε, οπότε το CETA Plus είναι αυτό το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε και νομίζω ότι οι Μεξικάνοι το έχουν καταλάβει, ήμασταν απόλυτα σαφείς. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ουσιαστικό το θέμα και έχει να κάνει με το πώς νομοποιούμε την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική ευρύτερα. Να σας πω τώρα πως τουλάχιστον για το πολιτικό σκέλος θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα αναστολής συμφωνίας, δηλαδή σε περίπτωση που ε, θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις να έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας είπαν πως καμιά φορά είναι πραγματικά αποτρόπαιο το τι συμβαίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να το εντάξουμε όχι μόνο στο εμπορικό σκέλος συμφωνίας αλλά και στο πολιτικό. Και βεβαίως για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, την καταπολέμηση και πάταξη διαφθοράς να είναι στο εμπορικό κομμάτι, να ε, συνδυάζονται με κυρώσεις και να έχουμε όλο το μηχανισμό ο οποίος θα είναι στέρεος και θα συνδέεται άρρηκτα με, το, με τα υπόλοιπα σκέλη. Δεν μπορούμε με τεχνητό τρόπο τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα αποσπάσουμε από την εμπορική πολιτική, τουλάχιστον όχι στα πλαίσια τούτη συμφωνία. Θα μπορέσει να αποτελέσει μια συμφωνία μοντέλο για την εμπορική πολιτική του μέλλοντο και είναι, όπω σα είπα, αναπόφευκτο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά ζητήματα και το περιβάλλον στη χώρα αυτή δεν είναι δυνατόν να ε, αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή σε μία διάσταση τα εμπορικά ζητήματα και μετά με ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκέλος ε, ε, τα θέματα αυτά. Όχι, θα πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο σημείο 18. Αν θυμάστε το σημείο 17 έχει αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση γιατί ο συγητής έχει αρρωστήσει. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 18, στην άλλη άκρη του κόσμου, στο χώρο ΑΣΕΑΝ. Εν ώψη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μαλαισία. Και ε, εδώ αν θυμάστε, έγιναν και κάποιες συνομιλίες με άλλα κράτη-μέλη του ΑΣΕΑΝ και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για διάφορους λόγους και στο μεταξύ έχουμε συνάψει συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, όχι εμείς δηλαδή ως κοινοβούλιο, ακόμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία βρίσκεται ε, προς εξέταση στο δικαστήριο. Έχει ολοκληρωθεί η σύναψη συμφωνίας με το Βιετνάμ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ε, στο στάδιο της μετάφρασης και ε, νομικής εξέτασης των επιμέρους σημείων και συμφωνία με την Ταϊλάνδη, με τις Φιλιππίνες και με την Ινδονησία επίσης. Αυτό λοιπόν δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια εποχή με μεγάλη δυναμική. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φίλιπ Τιρέτ, για, ε, υπεύθυνο για τις χώρες της Νότιας και Νότια-Ανατολικής Ασίας, έτσι ώστε να μας ε, παρουσιάσει το πώς έχει η κατάσταση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τις ε, τρέχουσες εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, Μαλαισία, για την οποία θα σας μιλήσω σε λίγο. Ήδη ο Πρόεδρος είπε κάποια λόγια στην εισαγωγή του. Να σας ενημερώσω όμως πώς έχουν τα πράγματα με το χώρο ΑΣΕΑΝ. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να συναυθεί συμφωνία στο 2019. Υπάρχει μεγά... Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες ε, ΑΣΕΑΝ. Όμως ε, το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει συναυθεί συμφωνία, δεν σημαίνει ότι ε, είμαστε και στάσιμοι. Γίνονται πολλές ενέργειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε ε, στα πρόθυρα ολοκλήρωση συμφωνία με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Οι διαπραγματεύσει με την Ινδονησία και τι Φιλιππίνες συνεχίζονται. Με την Ταϊλάνδη όμω και με τη Μαλαισία έχουν ανασταλεί προ το παρόν οι διαπραγματεύσει για ξεχωριστούς λόγους ε, στην περίπτωση τη κάθε χώρα. Υπάρχουν συζητήσεις με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και φυσικά εμείς συνεχίζουμε να, μην έχουμε, να έχουμε πρόσβαση χωρίς δασμούς στον χώρο ΑΣΕΑΝ. Είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία προστασίας των ε, επενδύσεων. Υπάρχει, λοιπόν, ε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα, γίνεται πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή στο χώρο ΑΣΕΑΝ και πρέπει να ε, σας πω επίσης ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, να υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ, αλλά προσπαθούμε να το, ε, να την διαμορφώσουμε ε, με συγκεκριμένα στάδια, σε συγκεκριμένα στάδια. Προσπαθούμε δηλαδή να αντλήσουμε έμπνευση από τις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν, τη συμφωνία ε, TPP για παράδειγμα, η οποία έχει διαφορετικές διατάξεις και δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία ως ένα παράδειγμα του πώς θα μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε την ε, δική μας συμφωνία. Μετά, η Επίτροπος Μάλιμστρομ θα δώσει μία ε, παρουσίαση, μία συνέντευξη όταν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Μανίλα με τους εκπροσώπους ΑΣΕΑΝ και θα γίνει επίσης και η διαβούλευση με τους Υπουργούς Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα. Όμως θεωρούμε πως ε, δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται να υπάρχει μία ε, κρίσιμη μάζα. Και εδώ θα έρθω στη Μαλαισία. Η Ζητήθηκε από τη Μαλαισία να ανασταλούν οι διαπραγματεύσει το 2012 λόγω των επικείμενων τότε εκλογών. Από τότε η Μαλαισία έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις διαπραγματεύσει για τη συμφωνία TPP, στην οποία προσχώρησε το 2010. και η ολοκλήρωση της συμφωνίας έγινε, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ήταν αρκετά ικανοποιητικά για τη Μαλαισία. Στο μεταξύ όμως η ε, Μαλαισία ε, λόγω της, ε, του, της κατάστασης του εισοδήματος έχει χάσει ε, το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων. Και αυτή τη στιγμή που η συμφωνία TPP βρίσκεται σε αβέβαιο στάδιο, η Μαλαισία έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Ανταγωνισμό μεταξύ άλλων από το Βιετνάμ και από άλλες χώρες. Μας βλέπουν με κάποια καχυποψία, ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που διαπραγματευόμαστε με, τον ανταγωνιστή της Μαλαισίας, την Ινδονησία. Μετά, να πω πως ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πότε θα ε, ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να είμαστε σίγουροι για το τι θέλουμε, ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Πρέπει λοιπόν να μην γίνουν λάθη και να διασφαλιστεί ότι η Μαλαισία όχι μόνο θα μπορέσει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε τι διαπραγματεύσει το 2012, αλλά να αναγνωρίσουμε και το γεγονό ότι έχουν αλλάξει οι πολιτικές μα σε ορισμένου τομεί. για παράδειγμα ε, για τις πρώτε ύλε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το εμπόριο ε, ορισμένων ε, πρώτων υλών. Και θα επιθυμούσαμε επίσης η Μαλαισία να προχωρήσει ακόμα περισσότερο σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα τη, τους όρους γεωγραφικής προέλευσης και της ε, δημόσιες προμήθειες. Τον τελευταίο χρόνο έγιναν διάφορες συναντήσεις, η τελευταία μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες με εκπροσώπους των διαπραγματευτών. Είδαμε ε, πως Υπάρχει μεν η καλή διάθεση από την πλευρά της Μαλαισίας να συνεχίσουν οι πραγματεύσεις, δεν έχουμε δει την στην πράξη κάτι τέτοιο, κάποια ε, τέτοια ε, προθυμία. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αρκετά λεπτή πολιτικά θέση, όμως ε, στις αρχές Μαρτίου στη Μανίλα ελπίζω πως θα λάβουμε τις πολιτικές διασφαλίσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουμε. Βέβαια να πω πως είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε ακριβώς την κατάσταση, είναι δύσκολο να υπάρξουν πολιτικές δεσμεύσεις, πόσο μάλλον όταν η οικονομία βρίσκεται ε, σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει όμως μία φιλοδοξία, ελπίζω αυτή η φιλοδοξία να είναι αντίστοιχη ε, της περίπτωσης ε, του Βιετνάμ. Και αυτό πιστεύω θα είναι ενδεικτικό και των υπόλοιπων διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες της περιοχής. 10 Μαρτίου λοιπόν θα γίνει η επόμενη συνάντηση και με την πρώτη ευκαιρία θα χαρώ να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα. Ε, τώρα επικεντρώθηκα στη Μαλαισία, βέβαια με τα χαράς να απαντήσω και ερωτήσεις για τις άλλες χώρες με τις οποίες έγιναν διαπραγματεύσεις αλλά, τη, αλλά αύριο στην ομάδα παρακολούθησης θα έχω την ευκαιρία να σα δώσω και περισσότερες λεπτομέρειε. Ο κύριο Καμά, λοιπόν, ο οποίο είναι ο μόνιμο συγητής για τη Μαλαισία και μετά ο Τέβιτ Μάρτιν, που είναι ο μόνιμο εισηγητής για την ΑΖΕΑΝ 6 στην Σιγκαπούρη. Κύριε Καμάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να πω πω δεν φανταζόμουν πώ θα ξανασυζητήσουμε τη Μαλαισία. Νομίζω ότι το 2012 ο κύριος Καζάχα από τους φιλελεύθερους ήταν τότε ο εισηγητής όταν είχαμε προχωρήσει αναστολή, οπότε με μεγάλη χαρά ε, ε, βρίσκομαι πάλι εδώ για να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί σας. Η δική μας ομάδα πάντοτε καλωσόριζε την ελεύθερο εμπόριο όπου υπήρχε δυνατότητα, όπως επίσης και τις σχετικές συμφωνίες. Όμως στην πραγματικότητα, και το λέω αυτό επειδή προέρχομαι από τους ακαδημιακούς, από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, να σας πω πως δεν πρόκειται για καθαρά εμπορική συμφωνία. Είναι μια ε, προτιμησιακή συμφωνία, δεν ανοίγουμε μεν στους δε όλους μας τις αγορές. Όχι, το κάνουμε ανά ε, κλάδο με προτιμησιακά συστήματα. Να σας πω λοιπόν για ποιο λόγο είμαστε τόσο πολύ υπέρ αυτής της συμφωνίας. Καταρχήν, για τις χώρες ΑΖΕΑ, να σας πω πως η Μαλαισία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος εκεί και είναι πολύ βασικός παίκτη στη σταθερότητα της ε, περιοχής. 16% αύξηση είχαμε στις εισορές από τη και να σας πω στο 90% είναι βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης, οι άμεσες ευρωπαϊκές επενδύσεις είναι πάνω από 60 δις. Οπότε καταλαβαίνετε πως πρόκειται για μια συμφωνία η οποία, τουλάχιστον σε, απλά οικονομικ, σε απλούς οικονομικούς όρους είναι μια την οποία πρέπει να συνάψουμε. Επίσης, σύμφωνα και με το οικονομικό σχέδιο του 2010 που είχε παρουσιάσει η Μαλαισία για να γίνει μια χώρα υψηλού εισοδήματος μέχρι το 2020, να σας πω πως έχει αναλάβει δεσμεύσεις η ε, πολιτική τάξη της, ε, και οι κυβερνώντες της Μαλαισίας. Ε, αυτή τη στιγμή το πλήστον των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται είναι σε κλάδους που μπορεί να έχουμε και ευρωπαϊκές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια και να σας πω πως ε, γενικά έχουν πετύχει τους στόχους που έχουν θέσει στο οικονομικό σχέδιο αυτό το 2010. Τώρα, για το κατά πόσο μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα βασιζόμενη σε στοιχεία και όχι σε προκαταλήψεις που ενδεχομένω έχουμε, θα πρέπει να δούμε καταρχήν τι γίνεται με τα πρωτογενή δάση στην Μαλαισία. Δεν έχουν μειωθεί τα επίπεδα εκεί και σύμφωνα με τον ΟΗΕ εκεί είχαμε από μία αύξηση. Άρα δεν είναι καταστροφική κατάσταση ε, στους οποίους θα μας οδηγούσαν να πιστέψουμε κάποιοι εδώ. Και δεν είναι το ίδιο με άλλες χώρες όπου πραγματικά νομοποιείται κανείς να ανησυχεί για τα επίπεδα δάσωσης. Να σας πω πως υπάρχουν μικροκτηματίε στην Μαλαισία οι οποίοι ανησυχούν για ε, πολυεθνικές λευκές ε, δυτικές που ε, συνεργάζονται με λευκές ε, ε, δυτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις για να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρεί κανείς πως εδώ προχωράμε σε μια κίνηση λευκού νεοϊμπεριαλισμού ή απεικιοκρατισμού που θα πιέσει του Μαλαισιανού. Να σα πω πω το εθνικό επίπεδο φτώχεια ε, πριν από μέχρι μερικά χρόνια ήταν στο 49,93% και καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει πέσει πάρα πολύ με αποτέλεσμα να είναι πολύ ψηλή ακόμα η φτώχεια στη χώρα αλλά να φαίνεται πω υπάρχει μια σημαντική πτώση άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και κυρίω με την πρόσφατη νίκη που είχαμε στην ψηφοφορία για τη ΣΕΤΑ θα πρέπει να προχωρήσουμε και σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών. Όπω είπε και ο, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπή, θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Την τελευταία φορά άλλη συμφωνία γιατί είχαμε κάποια καθόδη θέματα. Ε, αμφότερη. Η Επίτροπος κυρία Μάστρουπ είπε πω το 2015 σε κάποια εκδήλωση κοινή επιχειρηματική με τη Μαλισσή πω αν ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει, πρέπει να είμαστε σίγουροι πω και οι δύο πλευρέ θέλουν να συμβιβαστούν. Δεν υπάρχει λόγο να ξανακολλήσουμε στα ίδια θέματα στα οποία είχαμε κολλήσει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν η ερώτηση μου είναι η εξή. Εσεί μιλήσατε πριν από δύο εβδομάδε για τα διάφορε επαφέ που έχετε, αλλά ποιε είναι οι αρχικέ σα εντυπώσει. Ξέρω πως η Επίτροπος θα συναντήσει τον ομόλογο της στη Μανίλα Πιστεύετε να έχουμε κάποια διαφορά στην προσέγγιση που ακολουθούν, τουλάχιστον από τι αρχικέ εντυπώσει που έχετε, για εκείνα τα δύσκολα ζητήματα που είχαν προκύψει στο παρελθόν. Επίση, τι είναι διαφορετικό σήμερα Ξέρω πω ο Πρωθυπουργό είπε πω θέλει να ξεκινήσουν σύντομα οι συνομιλίες. Έχει την πολιτική βούληση, φαίνεται αυτό. Και ίσω είναι νωρί για σας να απαντήσετε, αλλά πείτε μου, εσεί πού βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση έτσι ώστε να ξεκλειδώσουμε τα δύσκολα ζητήματα που δεν μα επέτρεψαν να συνάψουμε συμφωνία προηγουμένω. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δίδη Μάρτιν έχει το λόγο. Ε, θα μιλήσω και για τη Μαλαισία και για τη Σιγκαπούρη. Ο η κυρία Ροντρίγκη είναι σκιώδη ηγήτρια, αλλά δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει. Καταρχά, ένα γενικότερο σχόλιο εκ μέρου τη ομάδα μου για το ε, χώρο ΑΣΕΑΝ. Αποδεχόμαστε ότι είναι μια πολύ σημαντική περιοχή οικονομικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες ε, συνεργασίας και δραστηριοποίησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο αυτό. Από την άλλη όμως αντιλαμβανόμαστε απόλυτα και την ε, κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί και την ε, θέση που έχει η κοινωνία των πολιτών, η θέση η οποία επιδεινώνεται και δεν βελτιώνεται. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Ε, συγκεκριμένα, για την Μαλαισία η συνάδελφός μου θα ήθελε να τονίσει ότι Εάν θέλουμε να ε, ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία, πρέπει να τεθούν ορισμένες προϋποθέσεις, όχι μόνο για το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά για μια ε, αυστηρή βιώσιμη ανάπτυξη υποχρεωτική και με τους κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τις ε, διασφαλίσεις που χρειάζονται έτσι ώστε όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και οι εργαζόμενοι να προστατεύονται παρκώς. Τώρα, σε σχέση με το φινικέλαιο, ε, δεν νομίζω πως χρειάζεται να αναφερθεί συγκεκριμένα το φινικέλαιο. Θα μπορούσαμε εδώ να αντιγράψουμε το κείμενο από τη συμφωνία με το Βιετνάμ, που υπάρχει ένα κεφάλαιο ε, που αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα και πολύ ε, αυστηρά στην βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Τώρα, τις γεωγραφικές ενδείξεις. Νομίζω πως μπορούμε να ε, ακολουθήσουμε εδώ το παράδειγμα ε, της Σιγκαπούρης. Η Σιγκαπούρη έχει αποδεχτεί τις δικές μας απαιτήσει. Μπορούμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο και για τη Μαλαισία. Τώρα, Σιγκαπούρη. Νομίζω πως ε, η Σιγκαπούρη έχει δείξει ιδιαίτερη υπομονή με το ότι εμείς θέλαμε να εξετάσουμε τη συμφωνία με το δικαστήριο κτλ. Δείξαν λοιπόν πολύ μεγάλη υπομονή για όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και θέλω να πω προς την Επιτροπή ότι από τη στιγμή που αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα προσπαθήσουμε και εμείς να ε, ολοκληρώσουμε το δικό μας κομμάτι όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τώρα, δεδομένου του μεικτού χαρακτήρα της συμφωνίας, ε, έχει την πρόθεση η Επιτροπή να χωρίσει τη συμφωνία σε δύο μεγάλα μέρη για τις ε, μεικτές αρμοδιότητες και ε, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα πώς προβλέπονται τα πράγματα. Τώρα, Μιανμάρ. Καταλαβαίνω πως η συμφωνία αυτή είναι δυσανάλογα ευνοϊκότερη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά προς τη Μιανμάρ. Ε, να πω όμως ότι ήμουν μέλος της ε, Task Force της Καθηνάστων και το σκεπτικό πίσω από την Task Force που, στην οποία συμμετείχα ήταν ότι η Μιανμάρ δεν άνοιξε μόνο επενδυτικές ευκαιρίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για επενδύσεις που βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ε, δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων, κοινωνική ε, εταιρική ευθύνη κτλ. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν μαζί με την Εμπορική και Επενδυτική Συμφωνία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μέρος της συμφωνίας με την Κολομβία τον οδικό δηλαδή χάρτη, έναν τύπο οδικού χάρτη για τις υπεύθυνε επενδύσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ευρωπαϊκές ε, εταιρείες έτσι ώστε να γίνονται υπεύθυνε επενδύσεις. Τώρα, ε, για τα εργατικά δικαιώματα στη Μιανμάρ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο της συμφωνίας με τον Μπαγκλατές. Όμως πιστεύω πως δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο στις ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά να επεκταθούμε. Αυτά που ακούω από τους εκπροσώπους στη Μιανμάρ είναι ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι μεν ε, λειτουργούν και δραστηριοποιούνται με τρόπο υπεύθυνο ε, άμεσα αλλά αυτό, αυτή η υπευθυνότητα δεν χαρακτηρίζει και τις ε, σχέσεις τους με τους προμηθευτές. χρησιμοποιούν κακοπληρωμένους ε, εργάτες, ε, α, ε, ακατάλληλες πρακτικές και συνθήκες εργασίας. Τώρα θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά να ολοκληρώσω με τις Φιλιππίνες και να πω ότι πριν από ένα-δύο χρόνια ήμουν από εκείνους που πίεζε για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τις Φιλιππίνες. Όμως πρέπει να πω ότι ε, δεν θεωρώ πως αυτή η στιγμή είναι η κατάλληλη για να συνεχίσουν ή να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις με τις Φιλιππίνες. Δεν ε, αναφέρομαι μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα που βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά και στο ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ε, πηγε, βαδίζει πολύ γρήγορα προς τη δικτατορία. Υπάρχει η κατάρρευση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και νομίζω πως θα ήταν λάθος χρονική στιγμή να εισέλθουμε σε διαπραγματεύσεις με τις Φιλιππίνες. Πόσο μάλιστα όταν ο γερουσιαστής Ελίμα, ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της κυβέρνησης, έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει ε, κατηγορίες ε, οι οποίες ε, στόχο έχουν να αποκλείσουν την κάθε μορφή ε, αντιπολιτευτικής φωνής στις Φιλιππίνες. Επίσης ε, γίνονται ε, δολοφονίες οι οποίες επίσημα συνδέονται με εμπόρους ναρκωτικών, όμως στην ουσία πρόκειται για πολιτικού χαρακτήρα δολοφονία, δολοφονίες. Ευχαριστώ πολύ. Η Αν Μαρή Μινέρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω μεγάλο πρόβλημα με την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Θα πρέπει η εμπορική πολιτική να είναι αμοιβαίως υποφιλής και η, πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξυπηρετεί κυρίως τις πολυεθνικές. Ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε τους εργαζομένους, ούτε εξυπηρετεί τις χώρες που πολύ δύσκολα αντέχουν σε ανταγωνισμό από μεγάλες οικονομίες. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η εμπορική πολιτική που αναπτύσσουμε ωφελεί μόνο τις πολυεθνικές εταιρείες. Τον ε, Οκτώβριο του 2013 ε, είχαμε μια συμφωνία για την προστασία των επενδυτών. Οι χώρες ε, της Ασίας όμως είναι ακόμη αναπτυσσόμενες χώρες, δεν είναι ακόμη εύρυθμα λειτουργούσες δημοκρατίες, ούτε έχουν πολύ αναπτυγμένο το σύστημα των υπηρεσιών. Οπότε ένα τέτοιο σύστημα προστασίας επενδυτών απειλεί τη δημοκρατία στις χώρες αυτές και μικρές χώρες ε, που υφίστανται τις πιέσεις των επενδυτών γιατί χρειάζονται επενδύσει, ε, γίνονται έρμεα αυτών των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Ουσιαστικά ακόμη και το τελευταίο, το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων ε, δεν θα έχει αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη που χρειαζόμαστε στις επιλύσεις των επενδυτικών διαφορών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο αυστηρές απαιτήσει στα εθνικά νομικά συστήματα πριν ε, συνάπτουμε συμφωνίες με τέτοιε χώρες. Επίσης, ε, θα πρέπει να καλύπτουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις ε, συμφωνίες, γιατί ακόμη και οι ευρωπαϊκές εταιρείε δεν εξασφαλίζουν επαρκή προστασία των εργαζομένων. Έχουμε πρόβλημα το φινικέλαιο, με την κλωστή φαντουργία σε χώρες όπω η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, ε, το φινικέλο στη Μαλαισία. Θα πρέπει λοιπόν να περιλάβουμε στι εμπορικές συμφωνίες και κάποιες διατάξεις που θα εξασφαλίζουν αηφόρο ανάπτυξη. Και στα πλαίσια τη συμφωνία με το Μιαμάρα ε, είμαι κατά τη συμπερίληψη του κεφαλαίου για τις επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά εδώ συζητάμε το ε, θέμα του STS, τη επιλύσης αφορών επενδυτή και κράτους. Ίσως πρέπει να ζυγίσουμε διαφορετικά τα πράγματα. Δέκα περιπτώσεις πέρυσι προσφυγής αυτό είχαν να κάνουν με ενέργεια και αυτές οι προσφυγές δεν ήταν από μεγάλες επιχειρήσεις αλλά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν αυτό το μέσο έτσι ώστε να δικαιωθούν. Γι' αυτό αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να ανανεώσουμε την ε, ενεργειακή χάρτα. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η Χέιτι τα έχει το λέγω τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αναφίβολο πως η απόρριψη της συμφωνίας του ειρηνικού, της εταιρική σχέση του ειρηνικού από τον πρόεδρο Τραμπ δίνει μια μοναδική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει πραγματικά ισχυρές, αναρρέ εμπορικέ συμφωνίε με τι χώρε ΑΣΕΑΝ. Και πιστεύω ότι έχουμε μια σημαντική ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ότι μέσω αυτών των εμπορικών συμφωνιών θα διαφυλάξουμε προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας, εργασιακών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα υψηλές προδιαγραφές. Ε, κάτι που σε κάποιο βαθμό θα ίσχυε και για την ε, εταιρική σχέση του ειρηνικού. Θα πρέπει λοιπόν να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Αναφερθήκατε κύριε Κεμάλ στο θέμα του Φινικέλαιου δεν είναι περισσότερο τώρα θέμα κάποιων κακών περιβαλλοντικών ομάδων που κατηγορούν τη Μαλαισία και την Ινδονησία για την καταστροφή και αποψήλωση των τροπικών δασών τους. Τώρα το παλάκι βρίσκεται στις ε, εταιρείε. Αυτές ζητούν κάποιες προδιαγραφές, όπως επισήμανε και ο κύριος Μάρτιν. ίδιες οι εταιρείε βρέθηκα επί τόπου και διαπίστωσα ότι κάποιε διεθνεί εταιρείε ε, πραγματοποιούν πολύ υπεύθυνε επενδύσει και μάλιστα μερικέ φορέ ε, πλήττονται από ε, τι εταιρείε που έχουν χαμηλότερε προδιαγραφέ ό,τι αφορά τι δοσοληψίε του με γηγενεί πληθυσμούς σε θέματα περιβαλλοντικά τουλάχιστον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η σχετική συμφωνία θα πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μια υπεύθυνη παραγωγή φινικελαίου και να περιλάβουμε και αυτό το προαιρετικό σύστημα μεν, αλλά δεν είναι ακόμη τέλειο. Θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη και αυτό το εθελοντικό σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, σε πολλές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητούμε εκθέσεις για το φινικέλο. Εγώ έχω την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι οι καλύτερες πραγματικά εταιρείε αναζητούν τρόπους ε, για διαφανή και ε, βιώσιμη παραγωγή, υπεύθυνη παραγωγή φινικελαίου. Διαρωτώ με λοιπόν αν θα λάβει υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σίγουρα υπάρχει το θέμα της αποψήλωσης των δασών και έχουμε λόμπι που συνδέεται κυρίως με την παραγωγή φινικελαίου στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς ε, με μηχανισμούς όπως το FLICT για τη διαχείριση των δασών ε, ή πώς μπορούμε να επενδύσουμε σε μια νέα διαδικασία καταπολέμησης αποψήλωση των δασών, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα την ε, Νοτιοανατολική Ασία. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε διάφορους μηχανισμούς και μέσα για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και ελπίζω να ε, λύσει τις απορίες μου σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, για τη Μιανμάρ, θεωρώ ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό και ως προς τον έλεγχο του στρατού ε, στους φυσικούς πόρους. Γι' αυτό και θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις αδιαφανείς δομές που ισχύουν στη Μιαμάρ και που δυσκολεύουν ε, τις, ε, τις ενέργειες, τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών εταιριών σε αυτές τις χώρες. Ευρωπαϊκή... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μία σειρά από ερωτήσεις που ακούστηκαν κυρίως για το θέμα της Μιανμάρ αλλά και για τη Μαλαισία όπως και για κάποιες άλλες χώρες. Στην πρώτη ερώτηση που έγινε για το κατά πόσο υπάρχουν ε, ε, ε, πεφρασμένες διαφορές με το πώς είχε η κατάσταση όταν ε, σταματήσαμε τις διαπραγματεύσεις το 2012, να σας πω ότι στη διαδικασία απογραφής σε κάποια σημεία οι Μαλισιανοί ε, έχουν μπει σε διάθεση διαπραγματευτική. Δηλαδή μας λένε θα το συζητήσουμε, ε, θα το συζητήσουμε αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις. Οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, αλλά μας προσφέρουν αυτές τις ε, δηλώσεις και βέβαια ε, ότι αυτό είναι σίγουρο θα φανεί μόνο όταν σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο συναντηθούμε για να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουμε αλλάξει σε σχέση με το 2012. Ε, Τώρα, έχει μπει στα πλαίσια της δια ειρηνικής συνεργασίας, δηλαδή με τις χώρες του ειρηνικού και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης εκεί και μπορούμε να δούμε τι έχει συμβεί ε, παρόλο που για το θέματα των δασμών και τα λοιπά, της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, εκκρεμούν κάποια στοιχεία. Ε, πιστεύω όμως πως παρόλα αυτά θα μπορέσουμε και εμείς να τρέψουμε το πλεονέκτημα των όσων έκανε και σε εσωτερικό επίπεδο η Μαλαισία για να ξεπεράσει κάποιους ε, θεσμικούς περιορισμούς. Κρατικές προμήθειες, για παράδειγμα. Εδώ ε, ήταν πάντα επίμαχο το θέμα, ποτέ δεν το είχε διαπραγματευτεί η Μαλαισία. Έχουμε κάποια έγγραφα αναφορά που κυκλοφορούν και θα θέλαμε να πάει λίγο πιο μακριά η Μαλαισία στο θέμα αυτό. Αλλά βέβαια έχουμε μόνο το αποτέλεσμα μια πρώτη διαπραγμάτευση, οπότε προφανέστατα υπάρχουν στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε. Ό,τι είδαμε και στην TTIP, δηλαδή ακόμα ε, για τις περισσότερες πολιτικές μπούμι πούτρα έχουν κάπως στεγανοποιήσει τους χώρους αυτούς, ε, οπότε για τις επενδυτικές ευκαιρίες εκεί δεν ξέρω τι έχω να πω. Πάντως έχουμε κάποια ξεκάθαρη μετακίνηση σε σχέση με τις θέσεις του 2012. Για το φινικέλαιο Νομίζω ότι είναι ένα εμβληματικό προϊόν της Μαλαισίας όπως και της Ινδονησίας. Είναι το βασικό εξωγικό τους προϊόν, πολύ επιθετικά τα συμφέροντά τους και όταν λέω επιθετικά εννοώ θέλουν να μειώσουν τους ε, δασμούς, να απελευθερωθούν από δασμούς για τις εξαγωγές αυτές και περιέργως πώς και οι δύο χώρες ε, επιβάλλουν κάποιους εξαγωγικούς δισμούς σε αυτά τα ε, προϊόντα, οπότε και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη ζυγαριά. Όμως η βιωσιμότητα εκεί είναι ένα περίπλοκο θέμα. Έχει να κάνει με τη δασική διαχείριση, με την ετικετοθεσία, με τη σήμανση, γιατί στις χώρες αυτές δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης για μικροκτηματίες. Και η Μαλισσία και η Ινδονησία συνεργάζονται και μάλιστα να σας πω ότι η Ινδονησία έχει το στόχο να ακολουθήσει και ένα ε, σύστημα υποχρεωτικό ε, πιστοποιητικού βιώσιμου φινικελαίου μέχρι το 2020. Η Μαλαισία σχεδόν τα έχει καταφέρει έτσι ώστε να εφαρμόσει και αυτή ένα υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης που αντίθετα με τα όσα κάνουν ε, στον ιδιωτικό, τα ιδιωτικά πιστοποιητικά θα δίνει η μεγαλύτερη προσοχή στους μικροκτηματίες και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο της ε, χρηστής διαχείρισης για το φινικέλο. Προφανέστατα λοιπόν, εδώ έχουμε θέματα περίπλοκα, τα οποία όμως είναι στην ημερήσια διάταξη και για μένα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το ότι και η Ινδονησία και η Μαλαισία αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν έχουν κάθε βούληση να ακολουθήσουν ένα σύστημα βιώσιμης ε, ανάπτυξης πολύ φιλόδοξο, όχι μόνο για το φινικέλαιο, αλλά και οι δύο χώρες γνωρίζουν πως υπάρχει μια αρνητική αντιμετώπιση για το φινικέλαιο. Και στην Ευρώπη και αλλού. Οπότε γι' αυτό σίγουρα θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Ο Ντέβιτ Μάρτιν μας έκανε κάποιες ερωτήσεις ε, για τις ε, γεωγραφικές ονομασίες προστατευόμενες. Ε, ίσως με τη Μαλαισία να έχουμε ε, κάποιο εμπόδιο γιατί έχουμε μια επιστολή μεταξύ Μαλαισιανών και ΙΠΑ αλλά δεδομένου ότι η ΙΠΑ αποσύρθηκε από, το, από την συμφωνία TTP ε, καταπίπτει η επιστολή και νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Βιετνάμ. Μιλήσατε για τη Σιγκαπούρη. Με το Βιετνάμ έχουμε μια εξαιρετική συμφωνία και νομίζω το Βιετνάμ είναι και στην TTP και έχει και δική μας και συμφωνία με εμάς, οπότε προφανέστατα το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Νομίζω πως καλό θα ήταν να έχουμε εδώ επαρκή προστασία για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις της ευρωπαϊκής. Ίσως δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολα τα θέματα με τη Σιγκαπούρη και έχουμε μια συμφωνία η οποία γράφει πριν από χρόνια και η οποία αναβαθμίστηκε για να έχουμε ε, ε, επενδυτική προστασία και μετά είχαμε και μια ευρωπαϊκή δικαστική υπόθεση στην οποία αναμένουμε τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου ίσως το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Ελπίδα μας είναι ότι εφόσον έχουμε την σαφήνεια της δικαστικής γνωμοδότησης θα μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε πιο γρήγορα με τη συμφωνία και να την καταθέσουμε και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως ένα ζήτημα το οποίο τρέχει παράλληλα ή το οποίο θα γίνει εντωμεταξύ αναμένοντας και τη γνωμοδότηση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι η αναβάθμιση του 14 για την προστασία των επενδυτών η οποία πλέον δεν είναι ενημερωμένη μια και έχει αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξαναεξεταστεί. Οπότε έχουμε συμφωνήσει με τη Σιγκαπούρη πως ο πιο εύκολος τρόπος και πολιτικά ίσως ο πιο ε, ξεκάθαρος τρόπος είναι παρόλη τον αρχικό δισταγμό της Σιγκαπούρης είναι να ξανανοίξουμε τη συμφωνία και να αντικαταστήσουμε τις διατάξεις του 14 με νέες επικαιροποιημένε. Αυτό ελπίζω πως θα ξεκινήσει είτε μέσα στον επόμενο μήνα είτε μέσα στους επόμενους δύο μήνες για τη Μιανμάρ τώρα πιο συγκεκριμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πιο λεπτομερείς συζητήσεις στην ε, Επιτροπή Παρακολούθησης. Θα έχουμε και τον βασικό μας διαπραγματευτή, τον επικεφαλής, αύριο. Στόχο μας είναι να ε, βελτιώσουμε την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα με τον τρόπο αυτό να μεταφέρουμε και τι ευέλικτε πρακτικέ στη χώρα. Όχι μόνο στις εγκαταστάσεις που θα έχουν στη Μιανμάρ, αλλά και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Για τη Μιανμάρ και το τι γίνεται με την επίλυση επενδυτικών διαφορών, να σας πω πως δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στις ε, διατάξεις που έχουμε για την προστασία των επενδυτών στην Μιανμάρ, αλλά το κείμενο που έχουμε και το οποίο σύντομα νομίζω θα κλείσει, είναι πραγματικά πολύ προχωρημένο. Άρτιο θα έλεγα και νομίζω ευθυγραμμίζεται με τα όσα έχουμε και να σας πω πως είναι το κείμενο που είχαμε στη ΣΕΤΑ με τον Καναδά συν όλες τις επιπλέον ε, διευκρινήσεις και προόδους που είχαμε κατά τη διάρκεια έγκρισης της ε, ΣΕΤΑ. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι έχουμε πραγματικά ένα επίκαιρο, επίκαιρες διατάξεις εκεί και όχι ένα πεπαλαιωμένο σύστημα επίλυσης διαφορών. Σας ευχαριστώ πολύ και εδώ θα ολοκληρωθεί αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης. Θα έχετε βέβαια σίγουρα τη δυνατότητα να επανέλθετε για αυτά που συζητήσαμε στο μέλλον. Να περάσουμε όμως στο σημείο 19 που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νορβηγίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αφορά τέσσερα κράτη. Σήμερα όμως δεν θα συζητήσουμε τόσο πολύ το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, αλλά κάποια τυπικά ζητήματα. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν ε, αφορά άμεσα εμάς, όμως από την άλλη επηρεάζει άμεσα και βαθύτατα ε, τις ε, διοργανικές μας σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Πρόκειται για μία συμφωνία που έχει συνάψει μόνο Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επίτροπος Μάλιμστρομ αναφέρθηκε σε αυτή τη συμφωνία στην ακρόασή και αναφέρθηκε επανειλημμένα σε αυτό ε, στο, στα πλαίσια συζητήσεων για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Ε, δεσμεύσεις δηλαδή, αναφέρθηκε σε δεσμεύσεις ε, που αφορούσαν το ότι δεν θα γίνεται τίποτα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Αυτό όμως δεν έχει τηρηθεί. Και εδώ στην Επιτροπή έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε επί του περιεχομένου. Να συζητήσουμε δηλαδή αυτά τα σημεία που ήταν προβληματικά τα σημεία που ενόχλησαν. Το θέμα δηλαδή αυτό που αφορά την, ε, το άρθρο 218 της Συνθήκης της Λισαβόνας για, την, ε, για το δικαίωμα άμεσης και πλήρους ε, ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων οποιασδήποτε συμφωνίας. Αυτό αναφέρεται ρητά και σαφέστατα στη συνθήκη και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, κάποια σοβαρά προβλήματα, παραλήψεις, παρατυπίες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Μογκερίνη διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο ε, για μας αλλά και για όλο το ε, πλαίσιο των διοργανικών σχέσεων. Άρχισε λοιπόν η διαδικασία αυτή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Σλοβακίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον ε, Επίτροπο Χάν. Καταλήξαμε στο ότι δεν θα ολοκληρωθεί καμία συμφωνία προτού αυτή η διάταξη αναφερθεί ρητά στις συνθήκες. Και αναφερθήκαμε λοιπόν στην εφαρμογή του άρθρου 218. Θα το συζητήσουμε λοιπόν σήμερα με έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Κλώτ Μέρτεν, ο οποίος είναι τμήματάρχης για την Δυτική Ευρώπη. Πρωτού όμως του δώσω το λόγο, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Μπορέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που είχε την καλοσύνη να θέσει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση, όπως μας υπενθυμίσατε, είχε ξεκινήσει ήδη από τις 30 Ιουνίου του 2016, παρουσία των πρεσβευτών της ε, Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Εκεί είπαμε τι ε, διαδικασία θα ακολουθήσουμε και συμφωνώ με την ακολουθητέα διαδικασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τώρα κάποια στοιχεία που αφορούν αυτή τη συμφωνία που εκπορεύεται από τη συμφωνία του ΕΟΧ του 1994 που μιλάει για τον νέο ευρωπαϊκό χώρο με τα, τα κράτη της ΕΖΕΣ και περιλαμβάνει και την Ορβηγία, Συλλανδία και Λιχτενστάιν. Η συμφωνία λοιπόν του 1994 επιτρέπει τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων εντός του ΕΟΧ χάρη στον χρηματοδοτικό μηχανισμό. Επίσης ε, και η Νορβηγία συνέβαλε ε, χάρη στο χρηματοδοτικό αυτό μηχανισμό, γιατί ισχύει για αυτήν ένας αυτοτελής ε, χρηματοδοτικός μηχανισμός και ο πλέον πρόσφατος χρηματοδοτικός μηχανισμός έληξε στις 30 Απριλίου του 2014, οπότε θα πρέπει να ανανεωθεί. Επίσης, με τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές ε, συζητήθηκαν και τα πρωτόκολλα για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Ορβηγία, ε, για την Αλία. Και επίσης τις συμφωνίες του 2015 καταλήξαμε σε συμφωνία και δύο πρωτόκολλα. Συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 και επίση συμφωνία με βάση τη χρηματοδότηση των πολιτικών συνοχή ε, εκ μέρου των χωρών ΕΖΕΣ και επίση συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου τη Νορβηγία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021. Και επίση πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και του Βασιλείου τη Νορβηγία και του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τη Ισλανδία. Τα δύο τελευταία πρωτόκολλα αφορούν την Ελία. Η Συμφωνία Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και η Συμφωνία της Νορβηγίας θα προβλέπουν από κοινού χρηματοδοτική συνεισφορά των ε, κρατών ΕΖΕΣ ε, του ΕΟΧ για την οικονομική και κοινωνική συνοχή ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2021. Με ε, αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη χρηματοδοτική ε, την αύξηση της ε, χρηματοδοτικής συμφοράς κατά 11,3% σε σύγκριση με την περίοδο 2009-2014. Στόχος είναι η φόρος ανάπτυξη και η λήψη υπόψη της ε, καινοτομίας, της έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, απασχόληση των νέων, κοινωνία των πολιτών και θεμελιώδη δικαιώματα. Μάλιστα η Ουγγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία και άλλες χώρες θα υποφεληθούν από την ε, συμφωνία αυτή. Και όπως μας υπενθύμησαν οι πρέσβεις ε, ε, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας τον Ιούνιο του 2016, ήταν πολύ φιλόδοξες αυτές οι προσπάθειες των χωρών ΕΖΕΣ και σημαντικές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος, επαναλαμβάνω, είναι ο περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά πρωτόκολλα για την αλληλεία, ε, μετά από ανάλυση των πρωτοκόλων προβλέφθηκαν νέε παραχωρήσεις προς τις χώρες αυτές για την περίοδο 2014-2021 με αύξηση των παραχωρήσεων και αδειών για κάποιες ε, δασμολογικές ε, ποσοστώσεις και για κάποιους γραμμές που αφορούν την δασμολογική ορολογία. Στην Επιτροπή μας θα εξετάσουμε και δύο συμφωνίες, αυτές με την Ισλανδία και την Νορβηγία. Οι διαπραγματεύσεις με την Νορβηγία έχουν ανασταλεί προς το παρόν παρά το άρθρο 19 της Συμφωνίας ΕΟΧ. Η αποδοχή των συνεισφορών των χωρών ΕΖΕΣ και της Νορβηγίας είναι κάτι πολύ θετικό και προβλέπει ε, συνεννόηση κυρίως σε θέματα γεωργίας ώστε να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να πληρώνουν τελωνιακούς δασμούς για ε, τυροκομικά προϊόντα και ε, κρέατα. Ελπίζω, παραλαμβάνω, να καταργηθούν επιτέλους αυτές, αυτοί οι δασμοί. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στις εμπορικές σχέσεις που θα έχουμε στο μέλλον και με την Ορβηγία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Κλοντ Μέρτεν από την Υπηρεσία Εξωτερική Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις και για το περιεχόμενο και για τις διατάξεις και βεβαίως και για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που έχουμε επιτύχει με τις χώρες ΕΖΕΣ και κυρίως για το χρηματοδοτικό μηχανισμό με την Ορβηγία για την περίοδο 14-21, όπως επίσης και με την επιπρόσθετο πρωτόκολλο ε, για την αλία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας. Οι εξελίξεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας που δίνουν την ευκαιρία στην Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο Λιχτενστάιν να χρησιμοποιήσουν τις τέσσερις ε, ελευθερίες της ε, ενιαίας αγοράς που βέβαια δημιουργούν όχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Ε, όπου πρέπει κανείς να ζυγίσει ποια είναι τα οικονομικά πλέον εκτίματα των χωρών ΕΖΕΣΑ από την συμμετοχή τους και από το πόσο μπορούν να ε, ευνοηθούν από την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή στην ενιαία αγορά. Εδώ ενισχύουμε τη συμφωνία του 1994, έχουμε βασιστεί στο άρθρο 115 όπου οι χώρες αυτές πάντοτε συμμετέχουν χρηματοδοτικά στην εξάλληψη των οικονομικών διαφορών που υπάρχουν στην, ε, στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Οπότε η Νορβηγία, όπως ξέρετε και εσείς, ήδη από το 2014 έχει συνάψει και έναν διμερή χρηματοδοτικό μηχανισμό, παρόμοιο με αυτό, μάλλον αυτό που μόλις ε, σας έχει παρουσιαστεί και πρέπει να σας πω πως το χρηματο... ο μηχανισμός ε, επιχορηγήσεων έχουν ήδη επικυρωθεί δύο φορές. Ο πιο πρόσφατος έληξε το 2014 και εν ώψη της συνεχιζόμενης ανάγκης να ελαφρυνθούν οι συνεχιζόμενες οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μέσα στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και πιο συγκεκριμένα μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 ξεκινήσαμε εμείς στην, εξωτερική, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα φιλόδοξο σχέδιο διαπραγματεύσεων έτσι ώστε αυτές οι επιχορηγήσεις να αυξηθούν, όχι μόνο να συνεχιστούν μετά το 2014, με αποτέλεσμα στις 3 Μαΐου του 2016 να υπογράψουμε τις σχετικές συμφωνίες οι οποίες προσωρινά έχουν εφαρμοστεί από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2016 και αποδεικνύουν πως υπάρχει βούληση από τις χώρες αυτές να ξεκινήσουν αμέσως ε, τις ε, διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΕΖΕΣ για τα διμερή μνημόνια ε, συνεννόησης, για τις κλαδικές προτεραιότητες, όπως επίσης και για την οικονομική εφαρμογή. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το πακέτο τεσσάρων συμφωνιών, το πιο σημαντικό είναι ο χρηματοδοτικός ε, μηχανισμός με την Νορβηγία, οι επιχορηγήσεις και οι ε, μηχανισμοί επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και πρέπει να σας πω πώς βασιζόμενοι στην προσωρινή εφαρμογή με κάποιες από τις ε, χώρες δικαιούχους έχουμε προχωρήσει αρκετά. Αναγνωρίζουμε πως αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός δημιουργεί δύο επιπλέον πρωτόκολλα για την Αλία με την Ορβηγία και με την Ισλανδία απορρέουν από αυτόν και έχουν ε, υπογραφεί παράλληλα ταυτόχρονα με αυτόν και επίσης βρίσκονται σε προσωρινή εφαρμογή και είμαστε ε, σίγουροι πως οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τους εμπλεκόμενους θεσμούς θα αποφύγουν τέτοιου είδου παρανοήσεις στο μέλλον σαν αυτές τις οποίες αναφερθήκατε εσείς. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας πρόθεση να προχωρήσουμε και να έχουμε μια κοινή κατανόηση για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε μελλοντικά. νομίζω ότι θα έχουμε μονογραφή και προσωρινή εφαρμογή αυτών των διεθνών συμφωνιών ε, σύντομα και παράλληλα θα έχουμε και την ε, συγκατάθεση του Κοινοβουλίου πριν την προσωρινή εφαρμογή. Αυτό είναι κομμάτι των ε, διαθεσμικών διαπραγματεύσεων και διοργανικών διαπραγματεύσεων και είμαστε πεπισμένοι πως και στο μέλλον οποιαδήποτε ενδεχόμενη παρανόηση θα αποφευθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο μόνος ηγητής μας, κύριος Πάμπριξ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσω με μια, ένα επικριτικό σχόλιο για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αξιοσέβαστη αυτή Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου. Αφενός, και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφετέρου. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που με προβληματίζουν, όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλούς άλλους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι επανειλημμένως ε, είχαμε καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα διεθνούς εμπορίου. Πρόσφατα μάλιστα κυρώσαμε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση ε, για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας δεν είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το πώς διεξήχθη η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σα φέρω μερικά παραδείγματα. Αναφερθήκατε ήδη στο θέμα Κατά βάση προσπαθούμε να δώσουμε μία μάχη και να διεκδικήσουμε το σεβασμό που δικαιούνται τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και πολλά εξαρτούνται από εμά. Αλλά η έλλειψη σεβασμού που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς ε, ε, δίνει βάσεις ε, σε μεταγενέστερες περιπτώσεις ώστε ε, σημαντικά θέματα εμπορίου να μην λαμβάνεται δεόντως υπόψη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη το καλοκαίρι στείλαμε επιστολή στην κυρία Μογκερίνη με πολλές ερωτήσεις για πολυάριθμε ζητήματα που άπτονται των σχέσεων της ε, Επιτροπής μας και της Νορβηγίας. Γιατί το δικό μας συμπέρασμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τα συμφέροντα των κρατών μελών και τα συμφέροντα των κοινωνιών μας δεόντως στις διαπραγματεύσεις που είχε με την Ορβηγία. Η απάντηση που λάβαμε σε ερωτήσεις μας και στην επιστολή του Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε βέβαια δύο μήνες μετά με κάποια καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, αργά παραποτέ. Αλλά πολύ λυπούμε που θα πω ότι δεν είμαστε ηλίθιοι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από εμά υπηρετήσαμε χρόνια ολόκληρα ε, στις κυβερνήσεις μας και ε, στέλνοντας μου μια απάντηση από την οποία δεν καταλαβαίνω τίποτα για, για τις ερωτήσεις που έθεσα, νομίζω ότι είναι περιττό να χάνετε το χρόνο σας στέλνοντα τόσο ακατανόητε απαντήσει. Καλύτερα να τον αξιοποιείτε καλύτερα από το να στέλνετε ε, δυσανάγνωστα ε, μηνύματα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από άποψη γραφειοκρατίας, ε, μερικέ φορέ φορές υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν ζητούμε κάποια θέματα μόνο και μόνο για τη χαρά της γραφειοκρατίας από καπρίτσιο. Απλώς ε, εδώ έχουμε διαφορετική άποψη της Νορβηγίας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διαφορά ε, τη, και την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πρόβλημα αλληλευτικό γιατί μία εταιρεία μας αντιμετωπίζει χρεοκοπία, βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης γιατί έχει επιβαρυνθεί από το νορβηγικό, νορβηγικό σύστημα και το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία πρωτοβουλία για να μας βοηθήσει. Μας λέτε ότι είναι ξεχωριστά αυτά τα θέματα. Όχι, δεν είναι καθόλου ξεχωριστά, γιατί εδώ μιλούμε για τις σχέσει ευρωπαικης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Νορβηγίας. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν και να είμαι σαφής. Πολύ φοβούμαι ότι έχει ε, δεν έχει γίνει σεβαστή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έδειξε έλλειψη σεβασμού όχι προ εμένα προσωπικά, αλλά προ την Επιτροπή μα, την ΙΝΤΑ και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί στέλνουμε σαφεί απαντήσει, ε, ερωτήσει, γνώμη, και απαντήσει ε, ακριβεί δεν λαμβάνουμε. Ερωτώ λοιπόν και τις άλλες εβδομάδες, άλλες ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πιστεύετε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σεβαστοί από τους πολίτες μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να αποφύγουμε ε, την ψηφοφορία για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας, να δώσουμε ένα μήνυμα με την ε, ενέργεια αυτή, ώστε αν θέλουμε μπορούμε να συζητήσουμε το ζήτημα στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Νομίζω ότι έτσι θα ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η πρότασή μου λοιπόν προ του συναδέλφου από τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Επίση, ζητώ από το Προεδρείο τη Επιτροπή να ζητήσει και προφορικές απαντήσεις ε, στην κοινοβουλευτική συζήτηση που γίνεται. Να δώσουμε προφορική ερώτηση και να απαιτήσουμε απαντήσεις και να στείλει τους αρμόδιους Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ικανοί να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε ασαφείς απαντήσει ε, ή από οικονομική ή από πολιτική άποψη και μάλιστα πολύ καθυστερημένα. Νομίζω ότι αυτό είναι το χρέο μα προ του ψηφοφόρου μα προ ε, τι χώρε μα, αλλά και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απαιτήσουμε αυτό το σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σαφέστατα το μήνυμα. David Μάρτιν, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήταν όντω σαφέ το μήνυμα και εγώ ελπίζω να είμαι σύντομο και εξίσου σαφή. Καταρχά, να είμαι ξεκάθαρο. Ελπίζω η ΕΕΔ να έχει την ίδια προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία προσωρινή εφαρμογή προτού δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ απόλυτα ε, σε όλα τα σημεία. Τώρα για την ε, ε, Νορβηγία, τη Γεωργία και την Αλία ξέρω ακόμα λιγότερα πράγματα, αλλά συμφωνώ ότι η Νορβηγία έχει σπάσει αυτό το καλό πνεύμα συνεργασία με την πράξη της. Καμία αντίρρηση. Τώρα, ε, εκεί που διαφέρω με, από τους συναδέλφους είναι ότι είναι στον ε, οικονομικό μηχανισμό της ΕΕΔ. Δεν θεωρώ πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλουμε την ατζέντα μας. Είναι δικά τους χρήματα, δεν είναι δικά μας χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε κάποιες από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νομίζω πως πρέπει να ε, εκβιάσουμε τις καταστάσεις στερώντας από αυτούς τους ανθρώπους κονδύλια που χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν ας ε, έχουμε αυτό υπόψη πρωτού ψηφίσουμε για ε, την οικονομική συνεισφορά. Σας ευχαριστώ. Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, λέει ο κύριος ε, Παλέσα, είναι ε, κάποιες ε, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αλίας στο, στα Σβάλμπαρτ και στο Σπίτσπεργεν. Υπάρχουν δικαιώματα πρόσβασης στους φυσικούς πόρους αυτού του αρχιπελάγους και αυτά διασφαλίζονται από τη συνθήκη του Σβάλμπαρτ όπως τη γνωρίζουμε συνθήκη των Παρισίων από, υπεγράφει από πολλέ μεγάλες ε, χώρες τη Ευρώπη την Πολωνία μεταξύ άλλων, τη Γερμανία, τις χώρες, τη Γαλλία. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί βλέπω μία ε, κατάφορη ε, παραβίαση των συμφωνιών, κατάχρηση των αλλιευτικών φυσικών πόρων τη περιοχή αυτή και βλέπω ότι η Νορβηγία δεν σέβεται τη συνθήκη των Παρισίων. Είμαι σίγουρος πως η, γνωρίζει τι συμβαίνει, γνωρίζει τι έχει κάνει η Νορβηγία. Πέρυσι το Δεκέμβριο μάλιστα είχε ε, δημοσιευτεί και μία σχετική ανακοίνωση από το υψηλότερο ε, επίπεδο της Ευρωπαϊκής Δίκης, το Συμβούλιο των Υπουργών. Έγιναν διάφορα, ε, έγινε δημόσια διαβούλευση και Είδαμε που καταλήξαμε. Μετά υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν, την, ε, έχουν εκδώσει άδειες αλίας και οι ε, πλειοκτήτες έκαναν επενδύσεις, προετοίμασαν, εξόπλησαν κατάλληλα τα αλλιευτικά σκάφη και δεν μπορούν να ε, αλλιεύσουν στα, στο αρχιπέλαγος αυτό. Όπως είπε και ο ε, συνάδελφος εισηγητής, υπήρχε νόμιμο δικαίωμα αλίας σε αυτήν την περιοχή. Παρόλα αυτά όμως ένα αλλιευτικό σκάφος ε, και ο διοκτήτης του συνελήφθη για παράνομη αλία, παρό, παρότι είχαμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να το κάνουμε. ως αποτέλεσμα αυτής της μονομερούς ενέργειας αυτής της τρίτης χώρας έχει σταματήσει η αλληλεία ε, από σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα είδατε αυτά. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω ποια είναι η επίσημη θέση της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εδώ. Πώς μπορούμε να επιτρέψουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ Τη Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι γίνεται με αυτήν την ε, απόλυτη έλλειψη σεβασμού ε, στις συμφωνίες από την Νορβηγία. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αγνοήσει τις επιθυμίες μας. Το 2013 εμείς ψηφίσαμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και να κάνει κάτι για αυτές τις ε, αυξημένες ε, τους ε, αυξημένους δασμούς. 270 αυξήσεις είχαμε και πρέπει να σας πω πως είχαμε στο Αρνί, στο Βόιο. Τίποτα δεν ήταν ασαφές για το ποια ήταν η θέση μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτές οι αυξήσεις της, ε, στους δασμούς είναι κατά του πνεύματος της συμφωνίας, είναι κατά του άρθρου 90, ήταν μονομερείς, προστατευτικές χωρίς να έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση. Εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε την εντολή να διαπραγματεύεστε εκ μέρους μας. Αλλά προφανέστατα δεν έχετε αναλάβει αυτή την ευθύνη με σοβαρότητα. Γιατί έχετε αγνοήσει τις δικές μας α, α, επιθυμίες και έχετε παραιτηθεί από τα διαπραγματευτικά μας ατού. Η συμφωνία αυτή της Νορβηγίας σε προσωρινό επίπεδο εφαρμόζεται και εσείς αγνοείτε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εμπορική πολιτική όπως περιγράφεται από τη συνθήκη. Και εμείς θεωρείτε πως η δική μας συγκατάθεση είναι απλώς διεκπεριωτική και δεν χρειάζεται να μας λάβετε υπόψη. Ε, η Θάτσερ μας είχε πει ε, κάποτε πως είμαστε κοινοβούλιο Μίκη Μάους. Ε, και εσείς ως θεματοφύλακας των συνθήκων μας φέρεστε σαν να είμαστε ε, Μίκη Μάους. Ε, τώρα κοινοβούλιο Μίκη Μάους. Οπότε στα 25 χρόνια που είμαι εδώ δεν είδα ποτέ τέτοιου είδους συμπεριφορά από κάποια εθνική κυβέρνηση ή διοίκηση. Και έχω τρεις σύντομε ερωτήσεις που θα ήθελα να μου απαντήσετε σήμερα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα γιατί αγνοήσατε τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Δύο αναγνωρίζετε εσείς τα λάθη των όσων κάνατε. Και τρίτον, τι θα κάνετε εσείς έτσι ώστε το σκάνδαλο αυτό να μην επαναληφθεί. Uh, Κύριε Ζιέρα, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι έκπληξη που σας ζητήσαμε να έρθετε, γιατί ζητήσατε να έχουμε προσωρινή εφαρμογή ε, αυτής της ε, συμφωνίας από το Συμβούλιο. Εμείς στις 5 Ιουλίου πέρσι ζητήσαμε να μην ζητήσετε να γίνει αυτή η προσωρινή εφαρμογή ε, των εμπορικών ε, κεφαλαίων των ε, συμφωνιών ε, σύνδεσης πριν τις εγκρίνει το Κοινοβούλιο. 5 Ιουλίου πέρσι. Οπότε τι σας εκπλήσει, γιατί σας καλέσαμε εδώ να μας το εξηγήσετε. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά μεγάλη έπληξη είναι πρώτα που παρόλα αυτές εσείς προχωρήσατε και δεύτερον πως χρειαστήκατε τόσο χρόνο μέχρι να έρθετε εδώ να μας δώσετε μια εξήγηση. Δηλαδή έχει φτάσει Μάρτιος πια για να ανταποκριθείτε σε ένα ουσιαστικό ερώτημα. τελείω τελείως απαράδεκτα και τα δύο. And that... Και εκτός από όλο αυτό, έχουμε και το εξή Δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Η Νορβηγία, όπως ακούσατε κι εσείς, το είπε ο συνάδελφος, αύξησε γεωργικούς δασμούς οι οποίοι... Να το πω διαφορετικά. Που ενδεχομένως είναι και κατά του γράμματος της συμφωνίας και σίγουρα κατά του πνεύματος της ίδιας συμφωνίας. Δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτή τη συμφωνία ε, με άλλο τρόπο. Είναι σίγουρο πως είναι κατά του πνεύματος όταν για το αρνί και το βόλιο έχει αυξήσει τους δασμούς. ίσως αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός είναι ένας τρόπος για να μας δωροδοκίσουν, για να ξεφύγουν από την παγίδα στην οποία έχουν υποπέσει και ίσως θα έπρεπε να τους αφήσουμε να το κάνουν. Αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Να το ψάξουμε. Όχι να αφήσουμε στην άκρη αυτή τη συζήτηση και να μας πείτε αυτό που θέλουμε είναι αυτό που αποφασίσαμε να το λύσουμε έτσι και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε και σας παρακαλώ πολύ. Απλώς διεκπαιρεώστε το. Δεν είναι εντάξει αυτό που μας ζητάτε. Αν τα κράτη-μέλη, και συμφωνώ με τον κύριο Παουλίξ, ας το, ας το κάνουμε για πρώτη φορά και α είναι το παράδειγμα. Εάν τα κράτη-μέλη θέλουν αυτά τα χρήματα, τότε βοηθήστε μα έτσι να υπάρχει τάξη στο πω λύνουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί α, με αυτόν τον τρόπο που έγινε δεν θέλω να ξαναγίνει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πω ήταν σαφέ το μήνυμα, κύριε Μέρτεν. Ε, εγώ ήμουν πιο διπλωματικός, έτσι, κατά τα εισαγωγικά μου σχόλια, αλλά οι συνάδελφοι νομίζω μίλησαν έξω από τα πόδια, ε, δόντια. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο σύστασης ε, σύντομα. Αυτό θα το συζητήσουμε και στους συντονιστές. Είναι όμως σαφές ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με αυτόν τον τρόπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα στείλουμε λοιπόν οπωσδήποτε μία επιστολή στην κυρία Μογκερίνη. Και καλό είναι πιστεύω να έχουμε αυτό το προηγούμενο, έτσι ώστε να πορευτούμε στις μελλοντικέ μας διαπραγματεύσεις για μελλοντικέ συμφωνίες. Θα θέλατε να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις ή όχι. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας ε, πληροφορήσω ότι σε αυτό το πακέτο των τεσσάρων συμφωνιών που διαπραγματευτήκαμε για το χρηματοδοτικό μηχανισμό και τα ληφτικά πρωτόκολλα, Φυσικά η ευθύνη των διαπραγματεύσεων του χρηματοδοτικού μηχανισμού εναπόκειται στην ΕΙΕΔ. Τα άλλα θέματα βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και Αλίας. Και ίσως ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, Θαλασσών που είναι παρόν θα μπορούσε να σας δώσει μερικά ζητη... μερικές απαντήσεις ε, για το, για το αρχιπέργο Σόλμπερτ και τα ληφτικά ζητήματα. Μάλιστα σήμερα γίνονται διαπραγματεύσεις ε, και για τη Γεωργία με την Ορβηγία. Γι' αυτό και απουσιάζουν ε, σήμερα εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά πολύ ευχαρίστως θα έρθουν σε μεταγενέστερη συνεδρίαση για να σας ενημερώσουν για την πορεία αυτών των διαπραγματεύσεων. Πάντως, ε, έγινε μία παρεξήγηση στο θέμα της προσωρινής εφαρμογής αυτών των τεσσάρων συμφωνιών. Πάντως, ε, το μήνυμα ελήφθη, το είπα και προηγουμένως, το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήφθη και Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον, ώστε η κοινοβουλευτική σας επιτροπή που έχει ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και το σχεδιασμό των εμπορικών συμφωνιών να, να συνεχίσει και στο μέλλον να διαδραματίζει το πολύ σημαντικό της ρόλο. Σας ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώσαμε το σημείο 19, δεν κάνω λάθος, ήταν της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει οι συντονιστές ε, να συζητήσουν ε, την ακολουθητέα πορεία στο ζήτημα αυτό. Και αυτό ήταν το τελευταίο θέμα μας πριν το μεσημερινό, μεσημεριανό διάλειμμα. Ραντεβού και πάλι στις 3 το απόγευμα. Καλή σας όρεξη.